στην καθήλυνα αρμόδια Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Σχόλια για την ημερήσια διάταξη παρακαλώ. Όχι. Α, για τα πρακτικά. Τα πρακτικά υιοθετούνται. Περνάμε στο πρώτο σημείο της ημερησίας διάταξης για σήμερα το απόγευμα.